και εξ ονόματος του Σκηνοβουλίου συγγνώμη για το ότι συνέβη τη Δευτέρα που μας πέρασε με διακοπή ρεύματο κλπ. και κυρίως ε, στους ε, διοικητικούς, στους θεσμικούς συνεργάτες που πάντα ερχόταν εδώ και που όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι εδώ υπέστησαν τα όσα συνέβησαν ε, και υποβάλλουν προτάσεις στις συντονιστές γιατί στο τέλος του πρωινού θα έχουμε μια συνάντηση των συντονιστών για να δούμε ακριβώς την ημερήσια διάταξη με την οποία δεν ασχοληθήκαμε είχαμε τη Δευτέρα να την διεκπαιρεώσουμε στο μέλλον. Εδώ τη Δευτέρα ακριβώς είχαμε κανονικά την εκλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής μας. Οι συντονιστές ε, θα το συζητήσουν αυτό το πράγμα γιατί θεωρούν ότι... Συγγνώμη το τηλεφωνό μου. Λοιπόν, οι συνθήκες ακριβώς ε, το ότι συμβαίνει γύρω από το πρόσωπο του νέου Προέδρου αξίζει να ασχοληθούμε μαζί ε, με το θέμα αυτό και να το συζητήσουμε. Για να ακούσετε τώρα και σε ποιες γλώσσες μπορείτε να μας ακούτε. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε πια βουλγαρικά, λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι για την, ε, τους ε, βούλγαρους βουλευτές μας γιατί χρειάστηκε να τους πάμε σε άλλη συνεδρίαση στην συνδιάσκεψη των Προέδρων. Αλλά έχουμε λιθουανικά, σουηδικά, ελληνικά, τσεχικά επιπλέον που δεν είχαν προβλεφθεί πριν. Κάτι ακόμα να σας υπενθυμίσω ότι ε, ηχογραφείται η συνάντησή μας αυτή και επίσης τον κύριο Κρίστιαν Ελέρς να καλωσορίσω που σαν διοικητικό υπάλληλο ε, μας έρχεται εδώ να τον χειροκροτήσουμε. Επίσης ας προσέξουμε κάτι. Ε, το πλευρά συναδέλφου Ήταλα έχει προταθεί για μέρος του λεκτικού συνεδρίου από την κυβέρνηση της χώρας. Ε, χειροκρότημα λοιπόν, είναι σημαντικές οι καινούριες του αρμοδιότητες και του εύχομαι να προωθηθεί όπως πρέπει. Είστε αξιόλογος ε, βουλευτής ακριβώς και είσαστε από τους καλύτερους εδώ και το να γίνετε μέρος του ελεκτικού συνεδρίου μας προκαλεί χαρά γιατί ας πούμε για ένας επίτροπος κάποιος απολεκτικό συνέδριο πρέπει να είναι πάντα από τους καλύτερους, από τους αριστούς μας. Ε, προχωράμε στην έγκριση της σημερινής διάταξης, της συνάντησης της 21ης Ιουνίου, καθώς και της 13ης, 14ης Ιουλίου. Σας έχουν ανακοίνωθει όλα αυτά και αν δεν υπάρχει μια κάποια αντίδραση, τότε μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα εγκριθούν οριστικά. Και όπως το έχουν ζητήσει αρκετά μέλη της Επιτροπής μας, ε, αναβάλλεται το σημείο 4 για τις 3 Οκτωβρίου για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων. Αυτό είναι το σημείο 4. Κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτό, όχι. Τίποτα. Όχι. Να προχωρήσουμε στο σημείο 5. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, την ημέσια διάταξη δεν εγκρίναμε, το λησμόνισα. Εντάξει, κάποιο αντίθετο με την ημέσια διάταξη, όχι, εγκρίνεται λοιπόν και η ημέσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 5, είναι σημαντικό αυτό το σημείο, είναι η μεταρρύθμιση τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά τη Απάτη. Ο Γενικός Διευθυντής όμως δυστυχώ ε, έχει καθυστερήσει, όχι όχι, εδώ είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη της ζητώ. Ο κ. Γκαλεά, το ελεκτικό συνέδριο. Όχι, συγγνώμη, από το δικαστήριο. Ingeborg Γκρέμπλε. Γκρέσλε. Με συγχωρείτε, ε, ναι, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε ναι, το σημείο 5. Μήπως θα ήθελες να μας παρουσιάσεις ε, τα πράγματα σχετικά με το θέμα αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη συζήτηση για τον για, τον, για την Όλαφ, τον, ε, τον κανονισμό 1073 σε 99. το Κοινοβούλιο λοιπόν το 2008 ενέκρινε τις νομοθετικές τροπολογίες με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Εν τω μεταξύ όμως η Επιτροπή ε, κατέθεσε τη δική της την ε, πρόταση η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών ε, αποφάσισαν ότι όσον αφορά αυτή την επεξεργασμένη πρόταση δεν θα πρέπει να καταθέσουμε νέα έκθεση αλλά εγώ να καταθέσω ένα έγγραφο εργασία και θα τοποθετηθούμε πάνω σε αυτή την ε, επεξεργασμένη πρόταση. Αυτό λοιπόν το έκανα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχετε μπροστά σας πέντε έγγραφα εργασία που προσπαθήσαμε να τα διατηρήσουμε σε έτσι διδακτικό ύφο, διότι θελήσαμε στους συναδέλφους ε, στο Κοινοβούλιο να δώσουμε την ευκαιρία να κατανοήσουν τι ακριβώς αποφασίσαμε το 2008. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα τέσσερα έγγραφα εργασίας ε, διαρθρώνονται γύρω από το δικαίωμα της ε, άμυνας και της εγγύησης προάσπισης κατά, κατόπιν ε, της μεθόδους έρευνας ε, τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, της ε, τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς και συντονισμός ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της απάτης, την καταπολέμηση της απάτης. Γύρω λοιπόν από αυτούς τους τομείς ε, το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει ήδη τις αρχικές του προτάσεις. Άρα δηλαδή εδώ βρισκόμαστε στην περίπτωση εκείνη όπου η υπηρεσία μετά από 10 χρόνια που ήδη υπάρχει πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος των προτάσεών μας. Ε, γύρω στις 100 τόσες τροπολογίες ε, καταθέσαμε. Έκανα λοιπόν το εξής. Έκανε αυτό που έκανε η Κομισιόν στην πρότασή της, στην αναθεωρημένη πρότασή της και πρέπει να σας πω, ε, δεν προσέθεσα τίποτα, ούτε αφαίρεσα, απλά τις αποφάσεις που έχουμε λάβει, τις ε, συμπεριλαμβάνω ε, και τις συνδυάζω σε σχέση με αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Βλέπετε λοιπόν, αν πάρετε τα έγγραφα εργασία και τα δείτε λιγάκι, και βεβαίως εδώ δεν μπορώ να σας διαβάσω το έγγραφο εργασίας και με λεπτομέρειες μάλιστα, όπως θα ήταν απαραίτητο ίσως, αλλά θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθεωρημένη πρότησή της ε, υιοθετεί μόνο εν μέρη τις δικές μας προτάσεις. Αυτό είναι νόμιμο. Όμως το πρόβλημα είναι ότι στην περίπτωση αυτή η Όλαφ ε, μόνο εν μέρη θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματά της. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ και επιμένω ως ε, στρατηγική διαπραγματεύσεων θα πρέπει να επιμείνουμε η Κομισιόν να υιοθετήσει περισσότερες δικές μας προτάσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, των εγγύσεων διαδικασιών και των ε, δικαιωμάτων των ατόμων που υπάγονται σε διαδικασίες διαδικασία Όλαφ. Ε, θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι παλαιότερα είχαμε μια ομάδα εργασίας διακομματική στην οποία συμμετείχε η Ίνες αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Σε αυτή λοιπόν την ομάδα εργασίας πραγματικά ε, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνένεση για τις ε, προτάσεις μας. Και στην αρχική πρόταση της Κομισιόν εγώ έχω καταθέσει 11 έγγραφα εργασία που σας καλώ να τα διαβάσετε. Εκεί λοιπόν εξετάζουμε τα προβλήματα αλλά και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα ε, πήραμε κάποιες αποφάσεις του Δικαστηρίου σε κάποιους τομείς και από αυτές τις αποφάσεις ε, προέκυψε ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Έκανα λοιπόν αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις και θέλω να σας πω ότι στη δική μου την ανάλυση όσον αφορά τις προτάσεις Κομισιόν το ερώτημα των εγγυήσεων για τις διαδικασίες και τα δικαιώματα της ε, υπεράσπισης, ε, αυτά δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά, που σημαίνει ότι στο σημείο αυτό πρέπει να επανέλθουμε. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή σε ορισμένους βασικούς ε, τομείς της αρχικής της πρότασης, τους τομείς αυτούς τους αναθεώρησε όσον αφορά παραδείγματος χάνει τον Review Advisor. Τότε το Κοινοβούλιο πρότεινε μια συγκεκριμένη διαδικασία και επίμεινε η διαδικασία αυτή να είναι ανεξάρτητη. Ε, θεωρώ λοιπόν επίση το εξή, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει για το σημείο αυτό ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας λέει και αυτή ακριβώ το ίδιο. Τώρα, οι δικές μας ε, οι διαπραγματεύσεις ε, αφορούν την Επιτροπή Εποπτείας ε, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε δύο βασικές μελέτες και των δύο οι μελέτες αυτές μας στηρίζουν ε, σε μεγάλο βαθμό και κατ' ουσίαν βλέπουν τα πράγματα όπως και εμείς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε κυρίως για ένα πράγμα. Εάν δεν εκμεταλλευτούμε την τρέχουσα μεταρρύθμιση για να λύσουμε τα προβλήματα της υπηρεσίας, τότε θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η Όλαφ θα παίρνει και άλλες αποφάσεις από το Λουξεμβούργο, ε, θα είναι όλο και πιο επίμαχο το όλο, η όλη κατάσταση η όλη διαδικασία και θα χάσουμε μια ευκαιρία να προωθήσουμε την Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Γι' αυτό λοιπόν στις επόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουμε να επιμείνουμε τα προβλήματα της Όλαφ ε, ως έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή ξεκινώντας από, την, ε, από το χρονικό διάστημα των διαδικασιών περνώντας τα θέματα της ε, εποπτείας αλλά και στα θέματα της υπεράσπισης. όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα επιλύσουμε. Διατυπώσαμε 14 ερωτήσεις ε, τις οποίες ε, καταθέσαμε και στους συντονιστές και λέμε ότι αυτές τις ερωτήσεις ε, πρέπει να τις υποβάλουμε και στο Συμβούλιο γιατί η ανατορημένη πρόταση δεν λύνει αυτά τα προβλήματα και η ανατορημένη πρόταση της Κομισιόν προσπαθεί αυτή την ειδική θέση της Κομισιόν που είναι διαθεσμικό όργανο που υπάγεται στην Κομισιόν, γιατί αυτή είναι η θέση της ε, Όλαφ. Ε, προσπαθούμε λοιπόν αυτό να το αλλάξουμε, κάτι που όμως ε, και το δεχόμαστε θα σημαίνει περικοπή των κοινοβουλευτικών μας δικαιωμάτων. Πρέπει βέβαια να το κουβεντιάσουμε, να δούμε τις παλαιότερες αποφάσεις. Νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη να διασφαλίσουμε την ε, λειτουργική ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Όλεφ. Και επίσης ε, έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις ε, απέναντι στους άμεσα εμπλεκόμενους να δημιουργήσουμε ξεκάθαρες δομές. Η Επιτροπή Επιπτίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αποτελεσματική εποπτεία γιατί για αυτήν την εποπτεία προβλέφθηκε εξάλλου. Στο Συμβούλιο υπάρχουν τώρα δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή λέει ότι αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει να κάνουμε τα λιγότερα δυνατά, αλλά κυρίως γρήγορα, με ταχύτητα. Και μετά να πάμε σε ενοποίηση των τριών νομικών ε, βάσεων. Και με βάση αυτές τις νομικές βάσεις να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της Όλαφ. Νομίζω λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά την εμπειρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η σχολή σκέψη δεν πρέπει επουδενή να υπερισχύσει. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι στην Όλαφ για μεγάλο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν με ασαφείς νομικές βάσεις, με επίμαχες νομικές βάσεις και αυτό ε, δεν πρέπει επουδενή να το επιτρέψουμε. Τη στιγμή μάλιστα που η ενοποίηση των νομικών βάσεων σίγουρα θα απαιτήσει τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια. Και σε αυτή την ενοποίηση των νομικών βάσεων αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι να διευκρινίσουμε τα δικαιώματα των κρατών μελών μέσα στην Όλαφ. Και ε, δεν πρέπει η Όλαφ να χάσει τα δικαιώματά της που έχει απέναντι στα κρατημέλη γιατί αυτά τα διεκδικήσαμε και αποκτήσαμε με πολύ κόπο. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω η μεταρρύθμιση που θα είναι μια μεταρρύθμιση μέσα στην ίδια την Όλαφ αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει με απόλυτη σοβαρότητα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και εμείς ως κοινοβούλιο ε, πρέπει να δεχτούμε ως βάση διαπραγμάτευσης αυτά τα έγγραφα εργασίας, τα οποία τι κάνουν τις παλαιότερες αποφάσεις του Κοινοβουλίου μέσω των κανονισμών, τα παρουσιάζουν, τα σταθμίζουν και επισημαίνουν που και πώς η Κομισιόν δέχτηκε θέσεις μας και ποιες απέριψε. Νομίζω ότι ε, θα είναι ενδιαφέρουσα η όλη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο θα την απολαύσουμε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι οι σκιώδεις ηγητές θα με στηρίξουν. Ε, θέλω επίσης να πιστεύω ότι στο μότο δυνατόν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε φιλική βέβαια ατμόσφαιρα, κάτι που πάντα ισχύει και συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιτύχουμε το μότο δυνατόν όσο το δυνατόν περισσότερες συναντήσεις. Πολλά θέματα πρέπει να επιληθούν σε τεχνικό επίπεδο. Ε, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα. Σε κάποια άλλα θα περιοριστούμε ή θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί συγκεκριμένων κειμένων πολύ νωρίτερα από ό,τι σε άλλα. Όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση της Όλαφ, εδώ υπάρχουν δύο δυνατότητες. Είτε το όλο θέμα θα αφαιθεί πλήρω στα χέρια του Γενικού Διευθυντή, άρα δηλαδή αυτό που αναφέρεται ω τα κείμενα θα πρέπει να διαγραφεί ή η δεύτερη λύση θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένη ενασχόληση σχετικά με τις εγγύησεις διαδικασιών, όπως το πρότεινε το Κοινοβούλιο αρχικά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Αυτά είναι τα θέματα όπου πρέπει να συμφωνήσουμε το στομότερο δυνατόν. Νομίζω λοιπόν ότι οι 14 ερωτήσεις που έχουμε διατυπώσει για το Συμβούλιο πρέπει να απαντηθούν προφορικά από το Συμβούλιο, γιατί αυτά θα είναι και τα ουσιώδη θέματα. Όσον αφορά λοιπόν ε, αυτό το έγγραφο εργασία που όπως σας είπα έχει ένα διδακτικό ύφος και προσανατολίζεται ε, και σε προβλήματα υπάρχει ένας πίνακας συνημένος με 120 σελίδες δυστυχώς μόνο στα αγγλικά και παρακαλώ να δείξετε κατανόηση σε αυτούς τους πίνακες βλέπουμε την αρχική πρόταση κομισιών, την αναθεωρημένη πρόταση της τις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Τροπολογία που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια και μετά στο τέλος την νέα ε, πρόταση Κομισιόν. Και άλλη μια ταμπέλα, ένας κατάλογος, όπου είναι τα δικά μου τα σχόλια. Και εκεί τοποθετούμε εγώ στις αλλαγές που έχει κάνει η Κομισιόν. Παρακαλώ να διανεμηθεί και αυτός ο πίνακας, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα της εργασίας ε, που έχει γίνει. Παρακαλώ λοιπόν να διανεμηθεί και αυτός ο πίνακας ε, των 120 σελίδων, γιατί είναι πολύ σημαντικός ε, και μπορεί κανείς να καταλάβει καλύτερα με τον πίνακα αυτό το κείμενο. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις ε, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Εποπτείας. Σήμερα θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να παρουσιαστούν αυτά τα κείμενα να μας εξηγηθούν. Ε, θα ήθελα να ε, λάβει το λόγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή Εποπτείας. Ε, ξέρω ότι ο αρμόδιος από την Επιτροπή Εποπτείας που πρόκειται να έρθει αρρώστησε, του εύχομαι καλή ανάρρωση, όμως θεωρώ ότι η άποψη της Επιτροπής Εποπτείας ε, πρέπει να παρουσιαστεί. Ίσως η γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας μπορεί να παρουσιάσει το, την ουσία. Η γνωμοδότηση είναι 17 σελίδων στα αγγλικά πάλι και δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό να μπορούν να το κατανοήσουν οι συνάδελφοί μας. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε ε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσα να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Εποπτείας για να μας εξηγήσει το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να λάβουν σοβαρά το θέμα γιατί ένα πράγμα είναι σαφές. Αν τώρα δεν καταστήσουμε αποτελεσματική την όλα αυτό θα είναι αδύνατον τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα ε, θα παρουσιαστεί αδράνεια και αυτό θα θέσει σε κίνδυνο και την ίδια την ύπαρξη της Όλαφ γιατί δεν θα είναι αποτελεσματική και δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που πραγματικά μαστίζουν αυτή την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα από την Επιτροπή μας να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, συγγνώμη και από τις υπόλοιπες ε, πολιτικές μάδες. Αλλά νομίζω ότι ε, ο αγώνας αυτός είναι, έχει πολύ περισσότερη σημασία από τη, τη μάχη κατά των λαθών ε, ενάντια στα λάθη, αλλά μας απασχολεί λοιπόν ιδιαίτερα. Έχουμε τα μέλη που περιμένουμε, αλλά δεν είναι ακόμα εδώ. Από το Συμβούλιο Εποπτείας λοιπόν της Όλεφ ε, θα θέλαμε να ακούσουμε τον κύριο με τη γραμματεία της με τη γραμματεία εποπτείας, ο κύριος Πετιγιών ε, που είναι παρόν. Μήπως κύριε Πετιγιών θα μπορούσατε να λάβετε τη λόγο για να μας παρουσιάσετε το θέμα, έτσι. Ναι, δέχεστε, δέχεστε. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι γιατί δεν έχω τη συνήθεια να παίρνω το λόγο σε τέτοιου είδους βήματα. Αντικαθιστώ τον κύριο Λόπες. Και άρα θα επαναλάβω απλώς τα συμπεράσματα <clears throat> της έκθεσής του που εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Και νομίζω θα έχει υποβληθεί αρμοδίως. Αν νομίζετε ότι μιλάω πολύ γρήγορα, <clears throat> να μου το πείτε για να το αλλάξω. Στις 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν εγκρίθηκε η γνωμοδότηση για την τροποποιημένη πρόταση που κατέθεσε η Κομισιόν στις 17 Μαρτίου. Η γνωμοδότηση αυτή ακολουθεί άλλες προηγούμενες του 2006 και του 2010 για την ανάλυση που είχε κάνει τότε η Κομισιόν. Η Επιτροπή Επιτήρησης έχει ξαναμιλήσει για τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν τα άτομα και που είχε κάνει η Όλαφ, τα πρόσωπα μάλλον. Αυτό όμως δεν το ξαναείπε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αντίθετα, αναφέρθηκαν άλλες λεπτομέρειες πρόσθετες καινούριε. Η Επιτροπή τονίζει ότι η Όλαφ είναι υπηρεσία έρευνας, διοικητικής έρευνας, για να προασπίζει τα συμφέροντα της Ένωσης και τις έρευνές της τις κάνει ανεξάρτητα. Διαπιστώσαμε ότι αντίθετα από το αρχικό κείμενο του 99, η μεταρρύθμιση που προτείνεται το 11 αφαιρεί από την Όλαφ κάθε περιθώριο ελιγμών ως προς την γνωστοποίηση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να επαναφερθεί αυτή η δυνατότητα γιατί είναι απαραίτητη για τις έρευνες. Γιατί επαναλαμβάνω είμαστε υπηρεσία ερευνών. Εφόσον λοιπόν στο βαθμό που η Επιτροπή μας βασίζεται στο σεβασμό των εγγύσεων που δίνονται για τα πρόσωπα πάντα λέγαμε ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στις τρέχουσες έρευνες. Εφόσον βέβαια υπάρχει εγγύηση της ανεξαρτησίας των ερευνών αυτών. Πράγμα το οποίο πρέπει να δηλώνεται ρητά στον κανονισμό. Οι έρευνες αρχίζουν με βάση γραπτές προσφυγές ή παράπονα. Πρέπει όμως η αίτηση να γίνεται επίσημα ή αυτεπαγγέλτος. Έτσι, δεν θέλουμε η έρευνα να γίνεται από το όργανο που αφορά το πρόβλημα, αλλά από ανεξάρτητο οργανισμό. Αυτό είναι σημαντικό και το λέει η γνωμοδότησή μας. Θεωρήσαμε επίσης ότι οι γνωμοδοτήσεις του Review Advisor δεν είναι της Όλαφ θέμα, γιατί έχει τη δυνατότητα να μην τις δεχτεί. Έτσι γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες και οι υπόλοιπε εγγυήσει που προβλέπονται, αλλά έτσι δεν χρειάζεται κάθε φορά να προσφεύγουν στον διαμεσολαβητή όσοι προσφεύγουν. Είναι και αυτό μια εγγύηση ανεξαρτησίας και πρόσβασης στους φακέλους της Όλαφ. Η τωρινή Επιτροπή Επιτήρησης αλλά και η προηγούμενη πρόσεξε ιδιαίτερα το θέμα της υποβολής πληροφοριών στις εθνικές αρχές. Με βάση την υπάρχουσα νομολογία θελήσαμε να διασφαλίσουμε την εγγύηση της, των πληροφοριών που δίνει η Όλαφ σε εθνικές δικαστικές αρχές. Αυτά με βάση τη νομική επιτροπή της Όλαφ που τα έχει συζητήσει επανειλημμένως αυτά τα θέματα και σε συνεννόηση με την Επιτροπή μας για την εγγύηση της βελτίωσης της ποιότητας των πληροφοριών αυτών που χορηγούνται. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί έτσι ώστε οι εθνικές διοκτικές αρχές να μπορούν σε περίπτωση απάτης να έχουν την καταλληλότερη πληροφόρηση. Ακούσαμε εμπειρογνώμονες και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αλλά και τονίσαμε ιδιαίτερα τη στιγμή της σημασίας που έχει η γνωμοδότηση ειδικών πριν χορηγηθούν οι πληροφορίες. Όποτε υπάρχει ποινικό αδίκημα θα θέλαμε να μην γίνεται συστηματική προσφυγή στις εθνικές δικαστικές αρχές και ορισμένες να την χάνουν απλώς διοικητικών κυρώσεων διότι μόνο οι εθνικές δικαστικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διατάξουν ή να μην διατάξουν την προώθηση ποινικών διώξεων. Καθήκον τους είναι λοιπόν της Όλαφ να συνεργάζονται πλήρως με τις εθνικές δικαστικές αρχές. Με σεβασμό βέβαια των ισχυουσών διαδικασιών έτσι ώστε τα μικρότερη σημασία αδικήματα να διεκπεραιώνονται ταχύτερα. Έτσι νομίζουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η απαραίτητη αυτή συνεργασία με τις Εθνικές Δικαστικές Αρχές. Τέλος, η Επιτροπή Επιτήρησης εκφράζει τη λύπη της γιατί το θέμα της πρόσβασης της Όλαφ σε όλες τις φάσεις τέτοιων ερευνών, ακόμη και την της πρώτης αποτίμησης, δεν έχει λυθεί ακόμη και θα θέλαμε ο κανονισμός να είναι από αυτούς αφέστερος. Η Επιτροπή μας ζήτησε την έναρξη διαλόγου με τις αρχές της Όλαφ εφόσον βέβαια αυτό δεν βλάπτει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η ανεξαρτησία του Γενικού Γραμματέα της Όλαφ και γι' αυτό δεχτήκαμε να το γράφει και στον κανονισμό. όλες οι πληροφορίες που προέρχονται από την Όλαφ είναι απαραίτητο να χορηγούνται στην Επιτροπή Επιτήρησης. Τέλος, με βάση αυτά που έγιναν λίγο μετά το θάνατο του κυρίου Μπρούνερ, προβλέπουμε την δημιουργία και μιας θέσης αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Αυτό είναι, αυτά είναι γενικά τα συμπεράσματα του κ. Λόπες που κανονικά θα έπρεπε να τα παρουσιάσει εκείνος σήμερα. Βέβαια θα είχε να προσθέσει μερικά σίγουρα αν ήταν εδώ, αλλά δεν είναι. Ευχαριστούμε για αυτή την πληρέστατη παρουσίαση. Ο δεν ήρθε ακόμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μήπως είναι εδώ ο τμήματάρχης του. κύριος Κέσλε είναι μαζί μας από την ΟΛΑΦ. Μπορεί να λάβει το λόγο λοιπόν για να ακούσουμε και την άποψή του. Με ιδιαίτερη χαρά μάλιστα. Κύριε Γενική Διευθυντή, συγγνώμη που δεν είπα ότι είστε παρόν ε, γιατί μίλησα πάντως για σας. Ε, είμαι ασυγχώρητος από τη στιγμή που δέχεστε λοιπόν ε, να λάβετε το λόγο κύριε Γενική Διευθυντά. Thank you very much, President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο λοιπόν. Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω αφού θα έχω ακούσει τις ε, παρατηρήσεις του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Όμως ε, είναι σαφές ότι ήδη μπορώ να πω, να μιλήσω, να πω πολλά. Υπάρχει τροφή σκέψης έχοντας ακούσει την άποψη της εισηγήτριας και την άποψη της Επιτροπής Εποπτείας. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να ισχυριστεί <laughs> ότι τουλάχιστον υπάρχει έλλειψη ε, προτάσεων, ε, ότι δεν έγιναν σκέψη κάθε άλλο. Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι δεν συμβαίνει αυτό συχνά, ότι για κάθε θέμα ε, αναλαμβάνονται ή εκδίδονται τόσο πολλές γνωμοδοτήσεις, δεν νομίζω, αλλά εδώ συνέβη και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι' αυτό. Δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες, διότι και εγώ κατά κάποιον τρόπο βρίσκομαι εδώ ως ε, παθητικός ε, ακροατής. Δεν είμαι εγώ εκείνος ε, που λαμβάνει τις αποφάσεις, αλλά είμαι εκείνος που θα κληθεί να εφαρμόσει αυτά που θα αποφασίσετε εσείς. Επειδή όμως μου ζητάτε τη γνώμη σας, θέλω και εγώ να πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής, η πρόταση του Συμβουλίου, ε, που είναι πολύ σωστά ε, διαρθρωμένες και γνωστές, και το έγγραφο εργασίας ε, του εισηγητή, του, της εισηγήτριας πιο συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτά μας επιτρέπουν ταχύτατα να προχωρήσουμε σε συμβασμό. Αν δεν θέλετε να μιλήσουμε για συμφωνία, ας πούμε σε συμβιβασμό. Γιατί βλέπω ότι οι προτάσεις αυτές ακολουθούν την ε, ίδια γραμμή. Ίσως ε, να υπάρχουν ε, κάποιες λεπτομέρειες για μικρότερα δευτερεύοντα θέματα, αλλά κατά την άποψή μου υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό για μένα, γιατί ανησυχούσα, φοβόμουνα και τους φόβους μου τους είχα εκφράσει σε αυτή την Επιτροπή. Ο φόβος μου λοιπόν ήταν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα υπάρχει ασάφεια σχετικά με την νομοθετική βάση, ε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινείται η Όλαφ. Αυτό βέβαια δεν, δεν θα βοηθούσε τις έρευνες που διεξάγει και σίγουρα δεν θα βοηθούσε και στο να ε, προστατευτούν ε, όσοι εμπλέκονται σε έρευνες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αμετάκλητο νομοθετικό πλαίσιο για τις ε, δραστηριότητες της Όλαφ και αυτό το χρειαζόμαστε ταχύτατα. Εγώ διάβασα όλες τις απόψεις που έχουν εκφραστεί και είμαι πεπισμένος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Και δεν είναι αυτό απλά ευσεβής πόθος. Είναι δυνατόν οι τρεις ε, θεσμοί και μέχρι το τέλος του έτους να αποφασίσουν. Βεβαίως και είναι παραμένει ευχή, αλλά είναι και μήνυμα, ένα μήνυμα που εκπέμπουμε από την Όλαφ. Το δεύτερο μήνυμα που θέλω να σας ε, αναφέρω είναι το εξής. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. να ακολουθήσετε το παράδειγμα των προηγούμενων νομοθετών. Αυτών δηλαδή που συνέταξαν τον ε, κανονισμό 1073 του 99, που βεβαίως και ο κανονισμός αυτός πρέπει να ε, επικαιροποιηθεί, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει εντωμεταξύ ο χάρτης δικαιωμάτων, αυτά έχουν αλλάξει. Αλλά ο κανονισμός 1073 ήταν ένα πολύ καλό νομοθέτημα και δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν σε ισχύ μέχρι τώρα απαράλλαχτος, χωρίς καμία τροποποίηση. Ένας λοιπόν από τους λόγους που συνέβη αυτό είναι ότι ο κανισμός 1073, ο κανονισμός αυτός δεν προέβλεπε υπερβολική έκδοση ρυθμίσεων για τα συγκεκριμένα θέματα που μας αφορούν. Βεβαίως τώρα όλα αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν, ε, πρέπει να ολοκληρωθούν, ε, πρέπει να προσθεθεί το θέμα των δικαιωμάτων ε, του ερευνόμενου, του κατηγορούμενου αν θέλετε. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε την έκδοση υπερβολικών ρυθμίσεων για την τελευταία λεπτομέρεια. Ε, για θέματα ε, λειτουργίας, ε, γραφείων. Να αποφύγουμε και την τελευταία λεπτομέρεια που θα αφορά στις έρευνες. Εσείς ίσως να διαφωνείτε, αλλά τα λέω όλα αυτά για τον εξή λόγο. Ο επόμενος κανονισμός μετά από αυτόν θα εκδοθεί και αυτός τουλάχιστον μετά από 10 χρόνια, το λιγότερο. Είναι λοιπόν μια δύσκολη, επίπονη, χρονοβόρα διαδικασία το να τροποποιεί ε, κανονισμούς. Ελπίζω λοιπόν ότι θα εκδώσετε ένα διαγωνισμό ο οποίος ε, θα είναι διαρκείας, θα αντέχει και βεβαίως και θα είναι και αποτελεσματικός. Ε, και αυτό μπορεί κανείς να το επιτύχει αποφεύγοντας, μόνο αποφεύγοντας υπερβολικές ρυθμίσεις σε οργανωτικά, διοικητικά θέματα και σε λεπτομέρειες. Πάντως, εκτός από κάποιες, όπως σας είπα, λεπτομέρειες, ο κίνδυνος ε, που περιέγραψα ε, δεν μοιάζει να υφίσταται. Ελέγχθησαν πάρα πολλά, συμφωνώ, ε, που ελέγχθησαν, ας πούμε, για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Ήδη ε, ζητήσαμε ε, να υπάρχει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για τα δικαιώματα των μαρτύρων, ε, των εναγωμένων, την ανεξαρτησία της υπηρεσίας, την ανάγκη η Επιτροπή Εποπτείας να ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από ε, την αρχή προστασίας ε, δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας ε, Δεδομένων από την Επιτροπή Εποπτείας, από τον Διαμεσολαβητή, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βεβαίως η λογοδοσία της Όλαφ η ανεξαρτησία, η ταχύτητα και η προστασία των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων, όλα αυτά είναι πολύτιμα και πρέπει να ε, βελτιωθούν, ε, πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχουν αντιφάσεις ε, μεταξύ αυτών όλων των στοιχείων. Άρα δηλαδή εδώ αυτό που τίθεται ως θέμα είναι να επικρατεί ισορροπία. Εγώ νομίζω ότι το κείμενο που έχει κατεθεί είναι ισόρροπο. Ορισμένες βέβαια προτάσεις της εισηγήτριας θεωρώ ότι επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να εξισορροπήσουμε τα αντικρουόμενα ε, συμφέροντα και απόψεις. Γιατί σας λέω, δεν είναι δυνατόν να βελτιώσουμε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν ε, την ίδια στιγμή και στην ίδια έκταση. Σας είπα ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά βεβαίως είμαι εδώ για να απαντήσω... Ε, στις ε, ερωτήσεις, αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να επισημάνω δύο πολύ σημαντικά θέματα επί της ουσίας. Το ένα θέμα είναι το θέμα που ετέθη πολύ σωστά από την εισηγήτρια και όχι μόνο από αυτή. Πρόκειται για τα δικαιώματα και για τις ε, διαδικαστικές εγγύησεις όλων εκείνων που εμπλέκονται σε έρευνες. Η τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν έχει ως στόχο να βελτιώσει και να διευκρινίσει τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Στην τροποποιημένη πρόταση προβλέπονται δικαιώματα, αυτά έχουν καταγραφεί, ε, προβλέπεται να ε, παγιωθούν μέσω της νομοθεσίας. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερωθεί, ε, να έχει δικαίωμα δικηγόρου. Συμφωνούμε επ' αυτών και ήδη και τα εφαρμόζουμε. Βεβαίω και αυτά πρέπει να κατοχυρωθούν νομοθετικά. Ήδη δηλαδή υπάρχει ε, μια σημαντική βελτίωση στην τροποποιημένη πρόταση. Ίσως να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά αν κατάλαβα καλά, η συγγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει και ο περίφημος review advisor όπως αναφέρθηκε. Δηλαδή, review advisor τι είναι, είναι κάποιος ο οποίος θα επιφορτιστεί στο να ε, εξετάζει διαμαρτυρίες του ενδιαφερόμενου. Αυτό υπάρχει ήδη όμως, υπάρχει και λειτουργεί. Τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες βέβαια, το θέμα είναι πώς θα οργανωθεί αυτό. Και αυτό προβλέπεται και στην τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν. Αν κατάλαβα καλά, η συγγήτρια προτιμά να υπάρχει διορισμός ενός ανθρώπου που θα ασχολείται με αυτό το θέμα αποκλειστικά και μόνο. Ένας υπάλληλο ο οποίος θα αναλάβει, όπως σας είπα, αυτή και μόνο την αρμοδιότητα. Ε, αυτό είναι οργανωτικής φύσης θέμα. Ε, τώρα, ε, κάθε φορά που χρειάζεται ένα ε, ένας υπάλληλο ανάλογα με την προϋπηρεσία του και τις ε, νομικές του γνώμης, γνώσεις επιφορτίζουν το να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτό πάντα κατά περίπτωση. Τώρα, αν Πιστεύετε εσείς ότι αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει σωστά μόνο αν υπάρχει ένας υπάλληλο ο οποίος θα έχει διοριστεί γι' αυτό και μόνο το θέμα και θα ασχολείται μόνο με αυτό, δεν ξέρω. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι επειδή θα έχει διοριστεί αντί να επιφορτίζεται κατά περίπτωση θα είναι πιο ανεξάρτητος. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι περισσότερο ανεξάρτητο ο άνθρωπο αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώ και αυτό θα διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή. Μπα περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αν τελικά συστήσουμε μια τέτοια υπηρεσία, γιατί ε, στην περίπτωση αυτή θα μιλάμε για ένα μόνο άτομο, θα έχει και τη γραμματέα του και άλλου συνεργάτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τίποτα σημαντικά. Το ότι υπάρχει ο θεσμό review advisor, αυτό είναι σημαντικό. Περιλαμβάνεται όμω ήδη στην αναθεωρημένη πρόταση. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί. Εμείς ήδη στην ε, εσωτερική μας ε, αναθεώρηση των ε, διαδικασιών της Όλαφ που ξεκινήσαμε, που δρομολογήσαμε το Μάρτι του προηγούμενου έτου μετά το διορισμό μου, ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση λειτουργίας της Όλαφ. Και ε, αναδιατυπώσαμε ε, τους εσωτερικούς ε, κανόνες. Και ήδη προβλέπουμε μία μονάδα, η οποία δεν θα υπάρχει σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες ερευνητικές μονάδες. Θα είναι μια άλλη μονάδα, την οποία θα απαρτίζουν νομομαθείς και η μονάδα αυτή, η υπηρεσία, το τμήμα αν θέλετε αυτό, θα ελέγξει, θα ελέγχει τη νομική υπόσταση περιπτώσεων κατά την έναρξη και κατά το κλείσιμο μιας έρευνας. Θα είναι λοιπόν ένα τμήμα το οποίο θα το αποκαλούμε Investigations Selection Unit. Δηλαδή θα είναι ένα τμήμα που θα επιλέγει ε, τις ε, ε, διαδικασίες και θα ερευνά όλα τα συμπαρομαρτούντα. οι όροι για τη σύσταση αυτού του τμήματος περιλαμβάνονται ήδη στην τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα όπου η τροποποιημένη πρόταση είναι τέλεια, γιατί λέει ότι ο Γενικός Διευθυντής πρέπει ε, να δέχεται συμβουλές επ' αυτού του θέματος και νομίζω η λειτουργία αυτού του τμήματος θα πρέπει να είναι υπό την αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή, όπως ήδη συμβαίνει βέβαια. Και πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία ε, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, ε, οργανώνουμε με την υπηρεσία μας για να μην δημιουργείται μια ακαμψία η οποία αν υπάρχει μας ε, δυσχεραίνει το έργο μας. Τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω, νομίζω ότι ήδη μακρηγόρησα, σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής Εποπτείας. Εσείς πρόκειται να συμβάλλετε κι εσείς στον ε, ορισμό αυτής της Επιτροπής Εποπτείας. Αν δείτε λιγάκι τις ε, δικές σας τις αποφάσεις για τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και αν τα συγκρίνετε αυτά με κάποιες από τις προϋποθέσεις που ήδη ισχύουν θα δείτε ότι υπάρχει αντίφαση. Δεν μπορεί η Επιτροπή Εποπτείας ε, να έχει μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες ε, μια συνάντηση εμπειρογνωμών δεν, δεν επιτρέπεται αυτό. Πρέπει λοιπόν να είστε πολύ προσεκτικοί. Να μην εκχωρήσετε στην, ε, να μην αναθέσετε στην Επιτροπή Επιπτίας κάποια καθήκοντα που εξορισμού δεν θα μπορούν να τα εκτελέσουν και ε, λόγω της πραγματικότητας δεν θα μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Παρεπιπτόντως, εγώ δεν βλέπω και την προστέμενη αξία του να υπάρχει άλλος ένας εξωτερικός οργανισμός ε, που θα συμμετέχει και αυτός στις έρευνες που διεξάγει η Όλαφ. Το τελευταίο που θέλω να πω για την Επιτροπή Εποπτείας αφορά ε, στο ρόλο της ε, στο φιλτράρισμα, στο πούμε, της ε, τελικής έκθεσης που στέλνει η Όλαφ στις εθνικές, στις εκάστοτε εθνικές δικαστικές αρχές. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Αυτό το ρόλο τον απέκτησε ε, η Όλαφ μετά από μια συγκεκριμένη περίπτωση που εκδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τώρα το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και ο νομοθέτης ε, καλείται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο ρόλος της ε, Επιτροπής Εποπτείας. Γιατί η απόφαση που ισχύει για την Επιτροπή Εποπτείας ε, είναι βέβαια νομολογία. Εγώ νομίζω όμως ότι η νομοθεσία υπερισχύει της νομολογίας, άρα δηλαδή και εσείς και εμείς δεν δεσμευόμεθα από μία απόφαση δικαστηρίου που και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ε, είναι λίγο και επίμαχη. Ε, εσείς βέβαια θα αποφασίσετε, αλλά δεν βλέπω την, τι αξία θα προσφέρει το να έχουμε μία Επιτροπή Εποπτείας η οποία θα έχει το, τη δυνατότητα να φιλτράρει περιπτώσεις που θα πρέπει να παραπεμφθούν στις εκάστοτε δικαστικές αρχές ή όχι. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι συναντιόνται μια φορά το μήνα η Επιτροπή Εποπτείας. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι μόνο αν συναντιόνται μια φορά το μήνα θα είναι αποτελεσματική. Μόνο τότε, ε, ίσως έχει νόημα αυτό που λέτε, ε, ίσως και να υπάρχουν και λάθη το να στείλει κανείς μια υπόθεση σε εθνικές δικαστικές αρχές, αλλά δεν είναι λάθος να στείλει κανείς μια παραπάνω υπόθεση, λάθος είναι ε, να στείλει κανείς μια λιγότερη υπόθεση. Πρέπει λοιπόν να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ε, αναθέσετε στην αρχή στην Επιτροπή Εποπτείας ε, ρόλους και καθήκοντα που δεν μπορούν να τα εκτελέσουν και που δεν θα προσφέρουν ε, αξία ε, στο σημαντικότατο ρόλο τους που είναι να μην επιλαμβάνονται κάθε φορά μεμονωμένων περιπτώσεων αλλά να καθιστούν την Όλαφ σε θέση, κατάσταση να μπορεί να λογοδοτήσει. Αυτά είχα να σας πω Πρόεδρο, και είμαι βεβαίω στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που ενδεχομένω θέλετε να θέσετε. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να εκφράσω ε, την ελπίδα μου ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μάλιστα σύντομα τουλάχιστον κατά διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης διαδικασίας. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Πολύτιμα τα στοιχεία που μας προσφέρετε και σας ευχαριστώ που μας τα κοινοποιείτε αυτά γιατί θα ξεκινήσει μια συζήτηση και από τη στιγμή που θα υποβληθούν ερωτήσεις σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε εκ των προτέρων να απαντήσετε. Πριν να ξεκινήσουμε την όλη συζήτηση, τώρα καλό να ακούσουμε και την άλλη άποψη γιατί την άποψη του δικαστηρίου, την προσέχουμε ιδιαίτερα, την ανεξάρτητη αυτή άποψη και Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου θα είναι σε λίγο. Δυστυχώς ε, υπάρχει πολύ πυκνή κίνηση, συμφόρηση, γι' αυτό καθυστέρησε. Ο κ. Μπετράγκουες μήπως θα μπορούσε να μας παρουσιάσει έτσι κάπως και εισαγωγικά την όλη έκθεση. Ο κ. Μπετράγκουες είναι στο τμήμα που ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό. Εντάξει, ναι. Ναι, Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, όπως το είπατε εσείς, αυτό το κείμενο του κύριου Γκαλέα, την εισήγησή του θα την κάνω εγώ. Πρώτα απ' όλα μας συγχωρείτε, αλλά δεν εξαρτάται από μας. Είναι στα αγγλικά το κείμενο του και γι' αυτό θα τα πω και εγώ στα αγγλικά. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να σχολιάσουμε την τροποποίηση της απόφασης της Κομισιόν για τις έρευνες της ΟΛΑΦ. Συμφωνούμε με τους στόχους της Κομισιόν στη μεταρρύθμιση αυτή. Την εξέβρεση δηλαδή μιας εξισορρόπησης μεταξύ ανεξαρτησίας και υπολογισμότητα. με αυτούς τους στόχους και εμείς κάναμε τις συστάσεις μας. Θα θυμάστε ότι δεν είναι η πρώτη προσπάθεια τέτοιας μεταρρύθμισης. Στην γνωμοδότηση 6 του 11 υπήρξε, υπήρξαν και προηγούμενες από το 2006 ήδη. Επίσης έγινε η ειδική έκθεση 2 του παρουσίασε το Μάιο ο κύριος Γκαλεάν όπου είχαμε τονίσει ιδιαίτερα τη σημασία της αποτελεσματικότητας των ερευνών της Όλαφ, δηλαδή πρέπει να επικεντρωθεί στα βασικά της καθήκοντα. Δεύτερον, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών της και τρίτον, η Επιτροπή Επιτήρησης να ενδυναμώσει την ανεξαρτησία της Όλαφ. Η απόφαση του δικαστηρίου ή του συνελεκτικού συνεδρίου που σας παρουσιάζουμε σήμερα τους ίδιους αυτούς στόχους έχει. Λοιπόν, εμείς τι διαπιστώσαμε. Ως προς τις τροποποιήσεις που προτείνονται, εμείς κάναμε μερικές παρατηρήσεις και σχόλια. Πρώτον, ότι η Κομισιόν δεν έκανε μία γενικευμένη πρόταση απλοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας κατά της απάτης. Δεύτερον, πρέπει να γίνει περισσότερο ανεξάρτητος έλεγχος, τρίτον να δοθεί περισσότερο βάρος στην προστασία των ε, δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τέταρτον, να διερευνηθούν παρατυπίες και σε μη χρηματικά θέματα του προσωπικού της όλα. Τέλος, να γίνει το κείμενο σαφέστερο και ευραχύτερο. Αναφέρουμε και συγκεκριμένα θέματα που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο για το μέλλον της Όλαφ. Τρία κυρίως. Πρώτον, ότι δυστυχώς δεν συνδυάστηκαν όλα τα νομοθετήματα που ισχύουν αυτή τη στιγμή κατά της απάτης. Και αυτό μας εκπλήσει. Γι' αυτό προτείναμε απλοποιημένη και συνδυασμένη νομοθεσία κατά των απατών και ζητήσαμε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν μια τέτοια πρόταση συνδυασμού. Δεύτερον, ο ανεξάρτητος έλεγχος του νόμιμου ή χαρακτήρα των ερευνών. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της μεταρρύθμισης. Ανεξάρτητος έλεγχος θα ήταν προς το συμφέρον και του ενδιαφερομένου, αλλά θα αύξανε και την νόμιμότητα της Όλαφ με περισσότερη χρησιμοποίηση της δυνατότητας να δοθεί χρόνος για να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους και οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό προτείνουμε να δημιουργηθεί η θέση του λεγόμενου review officer. Τρίτον, η διάρκεια των ερευνών. Εμείς πάντα λέγαμε ότι πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν ταχύτερα οι έρευνες και ταυτίσαμε στους προηγούμενους ελέγχους μας προβλήματα αποτελεσματικότητας και ταχύτητας διάρκειας των ερευνών. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει έκθεση και αναφορά η όλα κάθε εννέα μήνες. Εμείς ζητούμε δύο φορές το χρόνο. Ο στόχος να μειωθούν οι διάρκειες των ερευνών είναι βέβαια φιλόδοξος και γι' αυτό σχολιάσαμε την ειδική έκθεση της Κομισιόν, την πρώτη έκθεση για αυτό το θέμα από το 2005 ήδη και ζητήσαμε οι έρευνες να περιορίζονται ή δυνατόν σε έξι μήνες. Οι προτάσεις της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση είναι αξιόλογες, αλλά χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση αν θέλουμε να καταλήξουμε σε πιο αποτελεσματικό αντιαπατικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Αγιάλα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Γκρέσλε για όλη αυτή την εργασία, τις διευκρινήσεις της ε, και τις λεπτομέρειες της σχετικά με την όλη διαδικασία και ακριβώς ε, για να προετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση που θα είναι σχετικά με την έκθεση για τη μεταρρύθμιση. από τη στιγμή που πρόσεξα ιδιαίτερα και την πρόταση του, της συστάσης του ελεκτικού συνεδρίου, όπως επίσης και τις σημαντικές συστάσεις και διευκρινήσεις ακριβώς της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ, ο νέος Γενικός Διευθυντής που θα ήθελα να τον καλωσορίσω γιατί παραλαμβάνω τώρα ξεκινάμε σε μια σημαντική στιγμή για την όλη παγίωση του εγχειρήματο αυτού και για την αποτελεσματικότητα, την εξαρτησία να δούμε και να έχουμε την επόμενη μέρα ένα καλό σύστημα δικαστικό αστυνομικό και να λαμβάνουν υπόψη τους όπως πρέπει αυτή την εποπτεία, την παρατήρηση, τη μάχη κατά της απάτης εσωτερικής και εξωτερικής και σχετικά με ορισμένες ελλείψεις όμως ουσιαστικές. Λοιπόν, μετά από μια βαθιά ανάλυση όπως ακριβώς έχει γίνει με επαγγελματικό χαρακτήρα στην Όλαφ και για τα προβλήματά της φαίνεται και αυτό με ανησυχεί, φαίνονται μερικά στοιχεία που ήδη στο παρελθόν πολεμήσαμε εναντίον τους. Ο ρόλος της Επιτροπής Εποπτείας να μην κάνουμε λάθος στην περίπτωση αυτή. Αυτή η εγγύηση η ανεξαρτησίας, αξιοπιστίας της Όλαφ ε, σίγουρα περνάει μέσω της ανεξαρτησίας και της δυνατότητας για μια πολύ καλή, σωστή Επιτροπή Εποπτείας. Ε, επειδή το γνωρίσαμε ήδη, δυστυχώς, δυστυχώς ε, ήταν περίπλοκο το θέμα και έθεσε σε κίνδυνο άλλωστε στην συνέχιση της Όλαφ ε, έχετε και φίλους αλλά και αντιπάλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνω, κατανοώ την ειδική ευαισθησία που χαρακτηρίζει το θέμα και μετά από την ε, εξέταση αυτή λεπτομεριακά. Αλλά λόγω της πείρας ε, σας εγγυώμαι της ευρεία πείρα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή παρόμοια από οπτίε. Διαφορετικά θα έχει προβλήματα η Όλαφ. Βέβαια και πάλι σε τι επιμένουμε. Το καινούριο το σημείο είναι οι εγγυήσει των διαδικασιών να μην υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία και να εργάζεται επαγγελματικά η όλα φουδέτερα αντικειμενικά, επιστημονικά μπορούμε να πούμε και να αποφύγουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ή και υποψία γιατί ακούμε διάφορα πράγματα θα πρέπει όλα αυτά να αποτελούν μέρο τη διαφάνεια. θα πρέπει να λειτουργούν σωστά τα πράγματα, να μην υπάρχουν λοιπόν αμφιβολίε, να ξέρουμε κάθε φορά διάφανα ότι έχουμε ένα σωστό στο κατάλογο, ένα δεοντολογικό κώδικα μπορούμε να πούμε, για αυτές τις διαδικασίες ε, και τις εγγυήσει ε, και να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία που χρειάζεται η Όλαφ. Βέβαια, είχαμε πάντα πρόβλημα, το είπε και το ελεκτικό συνέδριο. Υπάρχει μια πρόκληση Παρακαλώ, θα πρέπει να το εξετάσετε, να το δείτε και θα πρέπει να βαστείτε και, στις βοήθειες, και στη βοήθειά μας. Υπάρχουν διάφορες προβλήματα σε διάφορα θέματα στα πλαίσια της Όλεφ εδώ και κάποια χρόνια. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορα κανθόδη θέματα, στα περισσότερα δεν είναι. Πρώτα απ' όλα οι προθεσμίες, ε, το πόσο γοργά προχωρούν τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια επιβράδυνση και αυτό είναι εις βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης. Αποτελεί λοιπόν ένα από τα προβλήματα και εμεί ακριβώς θα πρέπει να δούμε για την έρευνά μας, ε, για την ε, σχολεία της ΕΛΑΦ αυτά, να έχουμε ε, διάφορα παραδείγματα, διαδικασίες που να είναι υποδειγματικές και θετικές. Θα πρέπει μαζί να εργαστούμε και να ρίξουμε το βάρος μας για να μειώσουμε παρόμοια προβλήματα διαδικαστικά και να βοηθηθεί το προσωπικό επίσης και εσείς θέλετε να εργαστείτε σκληρά πραγματικά σχετικά με την εποπτεία αυτή και να μπορέσουμε επίσης να λύσουμε το θέμα της συνέχισης της διαφάνειας από τη στιγμή στιγμή που όλα αυτά προωθούνται και σε εθνικές αρχές, γιατί ε, διαφορετικά θα, έχουμε σε ένα, θα φτάσουμε σε ένα διέξοδο που θα έχουμε διάφορα θέματα που δεν θα μας διευκολύνουν και δεν θα έχουν μια καλή εικόνα της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν και πάλι σε επαναλάβω ότι έχετε την υποστήριξή μας για την ε, αυτή την εποπτεία και την εσωτερική και εσείς κυρία μου ναι, θα έχετε την υποστήριξή μας, είναι από τα σημαντικά θέματα αυτά και την υποστήριξή μας και η έκθεση αυτή να μην είναι απλά και μόνο λεπτομέρειες και λεπτομέρειες, να αποτελέσει ένα σημαντικό ευαίσθητο, ευέλικτο όργανο από τη στιγμή όμως που δεν αποδυναμώνεται ο τομέας των εγγύσεων και η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ εγγυάται τις δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις έρευνες, σε αυτή την εποπτεία, γιατί το είχαμε δει και στο παρελθόν ε, και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Ξέρουμε το παρελθόν τι έχει γίνει και ε, σίγουρα ε, ε, δεν θέλουμε να σας ενοχλεί το ότι τα προωθούμε αυτό. Θα πρέπει αντίθετα όλα αυτά να βοηθηθούν για να αυξηθεί η αξιοπιστία. Οι δυνατότητες λοιπόν της Επιτροπής Υποπτίας χωρίς καθυστερήσεις ε, γιατί δεν καθυστερεί τις υποθέσεις η Επιτροπή Απροπτίας, αλλά μπορέσει να επιταχύνει την όλη διαδικασία, την όλη κατάσταση και να μπορέσουμε όλοι μας να συνεργαστούμε μαζί της. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρέσλε. Ναι, ähm, Ο κύριος Γκάια. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, πρέπει να σας ε, ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Πρόεδρου μας, γιατί εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας είχε αναλάβει βέβαια να παρακολουθήσει αυτό το φάκελο ε, της κυρίας ε, Γκρέσλε. Αλλά και ο ίδιος ε, έγινε θύμα της διακοπής ρεύματος της Δευτέρας. Έπρεπε ήδη σήμερα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Μας ενημέρωσε πάντως για το πώς βλέπει αυτό το θέμα και ε, μας είπε ότι ε, σε πολλά σημεία στηρίζει την κυρία Γκρέσλε. Εγώ θα αναφέρω κάποιες ε, παρατηρήσεις, κάποιες ερωτήσεις. Πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις μου αφορούν στους παριστάμενους εμπειρογνώμονες και θα με ενδιέφερε να ακούσω τις ε, απόψεις τους, ε, τις απόψεις των διαφόρων θεσμών. Το πρώτο που θέλω να πω αφορά σε αυτή την πρόταση ενός αναπληρωτή γενικού διευθυντή. Ίσως να είναι ε, θέμα επιλογής λέξεων, αλλά στην έκθεση της Επιτροπής ε, Εποπτείας ε, διάβασα ότι αυτός ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής θα πρέπει να είναι της άμεσης εμπιστοσύνης της Επιτροπής Εποπτείας. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν είναι σωστό να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο αυτή η περίπτωση. Γιατί βρήκαμε ένα γενικό διευθυντή, πολύ κόπο και αυτό εκφράζει τη συνεργασία. Αν λοιπόν δεν ήταν θέμα σωστή διατύπωση, τότε διαρωτώ με γιατί στην Επιτροπή ενός αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως για τον ίδιο το Γενικό Διευθυντή. Ε, πρέπει να σας πω ότι από πλευρά νομιμοποίησης ε, δεν καταλαβαίνω. γνωρίζουμε ότι μέσα στην όλα ε, πολλές φορές υπάρχει διάσταση απόψεων και αν τώρα αυτό συμβεί και ανάμεσα στο Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή, ενώ και οι δύο έχουν νομιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εγώ σας εγγυώ με αυτόν τον τρόπο θα παραλύσει η Όλαφ. Και αυτό ε, σαφώ και δεν το θέλουμε. Όσον αφορά λοιπόν το ε, ρόλο και την επιλογή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή, επ' αυτού θα ήθελα να γίνει σε βάθο συζήτηση. Το δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω αφορά στην ε, αυτόματη ε, πρόσβαση στην ενημέρωση. Εδώ πρέπει να έχουμε ένα κανονισμό ε, που να είναι σε συμφωνία με, τον, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων. Πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε την άποψη του ε, επιτετραμένου με θέματα ε, προστασίας δεδομένων του Ευρωπαίου για τα θέματα αυτά. Τώρα, κάτι άλλο που έχει σχέση με το πώς αναφέρονται τα κράτη-μέλη, πώς καταθέσουν τις εκθέσεις τους, πώς θα συντάσσονται αυτές. Σήμερα έχουμε κάνει την εμπειρία ότι ε, τα κράτη-μέλη, όταν πρόκειται ε, για περιπτώσεις της Όλαφ, δεν κάνουν αυτό που θέλουμε. Πώς θέλουμε λοιπόν να αγγιηθούμε αυτή η αναγκαιότητα υποβολής εκθέσεων να καλύπτεται από τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκθέσεις, καταλαβαίνετε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε μια επιθυμία, να απευθύνουμε έκκληση, αυτό το στηρίζουμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε ε, να εγγυηθούμε την επιτυχία του εγχειρήματο. Και το τελευταίο μου ερώτημα αφορά στο θέμα της ε, μεταφοράς των αποφάσεων de minimis. Ε, το να εκχωρηθεί πάλι και αυτό στα κράτη-μέλη. Και διερωτώ με κατά πόσον η Όλαφ έχει τη δυνατότητα τη στιγμή που γίνονται περικοπές ε, στον προπλογισμό, διερωτώ με κατά πόσον η Όλεφ έχει το απαραίτητο προσωπικό, αν θέλετε, να εγγυηθεί κάτι τέτοιο και να, δίδεται, να δίδει τόσες πολλές ε, πληροφορίες ε, στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σέσκοβα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για όλη την πληροφόρηση που μας έδωσε. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τα καινούργια κράτη-μέλη. Χάρη στην πληροφόρηση αυτή και σε αυτά τα έγγραφα μπορέσαμε και εμείς να μάθουμε όλα αυτά τα θέματα και την ιστορία, το ιστορικό των προτάσεων. Έχω ορισμένα σχόλια. Πιστεύω ότι ο Review Advisor είναι κάτι που θα διευκολύνει κατά πολύ την εγγύηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσώπων. Είναι σωστό να υπάρχει μία ανεξάρτητη αρχή, ένας ανεξάρτητος αξιωματούχος για αυτό το θέμα ειδικά. Δεν συμφωνώ με τα συμπεράσματα της Κομισιόν ότι αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να αναλυφθεί από πολλά άτομα <clears throat> που ταυτόχρονα να ασκούν και άλλα καθήκοντα. Συμφωνούμε λοιπόν με τον εισηγητή ότι αυτό θα ήταν αντιφατικό, θα δημιουργούσε αντιφατικά συμφέροντα. Ένας ανεξάρτητος review advisor νομίζω ότι θα ήταν κάτι σωστότερο. Επίσης συμφωνώ με την πρόταση η Όλαφ για τις έρευνές της να πρέπει να χορηγεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Αλλά για τα διαμεθοριακά εγκλήματα και παρατυπίες δεν πρέπει η Όλαφ να δαπανά περισσότερα χρήματα για τέτοιες ποινικέ υποθέσεις που είναι δικαιοδοσία άλλων. Επίσης συμφωνώ να δημιουργηθούν σαφέστεροι κανόνες και πιο δεσμευτικοί για τις έρευνες. Η δημοσίευση όλων αυτών των κανονισμών όπως την προβλέπει η Κομισιόν δεν αρκεί πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός της διαφάνειας. Όσο για τις περιοδικές εκθέσεις, η εισηγήτρια στο τρίτο έγγραφο εργασίας της λέει και συμφωνώ ότι όπως λέει και η Κομισιόν η χορήγηση πληροφόρησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκεί να υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να κάνουν τακτική ενημέρωση της Όλαφ για ό,τι έχουν πράξει για μια έρευνα θα ήταν άχρηστο πρόσθετο βάρος για τα κράτη-μέλη και η Όλαφ επίσης θα επιβαρυνόταν γιατί έτσι θα χρειαζόταν να κάνει και αυτή η περιοδική αποτίμηση της πληροφόρηση που θα τις δίνουν πια τα κράτη-μέλη. Γκέσλερ. Και εγώ έχω μία ερώτηση προς το Γενικό Διευθυντή. <clears throat> Θα ήθελα να παρακαλέσω Όσον αφορά τον περίφημο Review Advisor, να μου εξηγήσετε γιατί η Κομισιόν το 2006 εφευρίσκει αυτό τον Review Advisor. Η Κομισιόν τον εφήβρε. Δεν τον εφήβρα εγώ, ούτε καν θα μπορούσα και να ήθελα. Δεν έχω την απαραίτητη φαντασία. Εφήβρε λοιπόν η Κομισιόν αυτό τον Review Advisor ε, και μετά από τέσσερα χρόνια θέλει τώρα να τον αποσύρει. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Τουλάχιστον όχι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όλοι να διρωτώνται τελικά τι γίνεται εδώ. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο ρόλο του Review Advisor. Και εγώ θα ήθελα να μας πείτε πώς ακριβώς άλλαξε ο ρόλος του Review Advisor μετά από τις διάφορες προτάσεις. Το ελεγκτικό συνέδριο πολύ σωστά μας υπενθύμησε ότι αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με την τέταρτη πρόταση της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση της όλα. Να επισημάνω λοιπόν, αυτό δεν ήταν δική μου ιδέα, ο Review Advisor, και να επισημάνω ότι αυτά που έχουν κατατεθεί και πάλι δεν είναι ικανοποιητικά. Η επανεξέταση των ε, διοικητικών ε, διαδικαστικών δικαιωμάτων. Ε, αυτό έχει τεθεί πιτάπιτος και τελικά αν θέλουμε από όλα αυτά να βγει κάποιο νόημα, δηλαδή ο review advisor να είναι κάτι που πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Εγώ ε, ποτέ δεν μου πολύ άρεσε ε, και με τον τότε Γενικό Διευθυντή το συζήτησα το θέμα. Δεν θα είναι τόσο απλά εφόσον έχουμε φεύγει αυτόν τον review advisor, δεν είναι απλό να τον αποσύρουμε, ε, γιατί ε, πλέον ε, έχει κάπως απλώσει τα πλοκάμια του και έχει καταξιωθεί κατά κάποιον περίοδο τρόπο και στο, στην άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. πρέπει λοιπόν να δούμε λιγάκι το θέμα των διοικητικών εγγυήσεων, διαδικαστικών εγγυήσεων. Εγώ τώρα, εν πάση το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν τον εφήβρα εγώ αυτό, το, αυτό το, το, αξίωμα. Και θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, τον Γενικό Διευθυντή. Βλέπω ότι θα κάνετε οργανωτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, καλό αυτό γιατί πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην Όλαφ. Βλέπω όμως ότι εφαρμόζεται ήδη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως προτρέχετε λιγάκι, γιατί ισχύει ακόμα στην απόφαση και έχουμε και εμείς λόγο. Ενδέχεται λοιπόν στο τέλος ε, εμείς να καταλήξουμε σε διαφορετική άποψη και πραγματικά εξεπλάγει για το ότι θελήσαμε να επιταχύνουμε την νομοθετική διαδικασία και να την επιβάλλουμε ίσως σε άλλους, σε εμά το Κοινοβούλιο. Άρα δηλαδή να καταγράψετε παρακαλώ στα πρακτικά ότι εγώ δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο. Δείτε το εξή ερώτημα ή θέμα και γι' αυτό αυτή η Review Procedure for Legality ε, με βάση αυτό πρέπει να δούμε η αποφάση της Όλαφ υιοθετούνται σε επίπεδο εθνικό ή όχι, μεταφέρονται εκεί. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, το ρόλο της Όλαφ για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και όσον αφορά την οργανωτική μεταρρύθμιση, θέλω να σας πω ότι όσον αφορά την αξία των ε, αποτελεσμάτων ερευνών, θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Γενικού Διευθυντού επ' αυτό. Και θέλω να πω ότι αυτή η ε, Επιτροπή Εποπτείας ε, πρέπει να ενισχυθεί ε, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγγυόμαστε τον εσωτερικό έλεγχο. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο προλαλής σας. Ε, και εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ε, δημιουργήσουμε έναν ε, αντίποδα. Νομίζω στον κατάλογο που σας ανέφερα προηγουμένως υπάρχει ένα σημείο όπου κάνω λόγο για τον απληρωτή γενικό διευθυντή. Λέμε εκεί ότι θέλουμε να ενημερωθούμε ποιος είναι, ποιος θα είναι αυτός και η Επιτροπή Εποπτείας θα πρέπει να μπορεί να τοποθετείται ε, στην επιλογή του αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε τελικά ποια διαδικασία θα επιλέξουμε. Και το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξή. Συναντήθηκα μία φορά με την Πολωνική Προεδρία και αυτό που βρίσκω καταπληκτικό στην Πολωνική Προεδρία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, θέλουν οπωσδήποτε να προχωρήσει το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως να μην ε, το καταλαβαίνετε, αλλά είμαστε σε μια ιστορική καμπή. Έχουμε μια Πολωνική Προεδρία που θέλει πάση θυσία να προχωρήσει ε, θέλει να συνεργαστεί πάση θυσία με τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν είναι ε, μια πολύ καλή είδηση για όλου μας και αυτή την ευκαιρία, την μοναδική και ιστορική που μας προσφέρεται, θέλουμε να την αδράξουμε. Ο Γενικός Διευθυντής έχει το λόγο. Euh, Θα θέλατε να λάβετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν. Αφού τα άκουσα όλα αυτά, αισθάνομαι μεγαλύτερη ανακούφιση. Θα σχολιάσω μερικά από αυτά που υπόθηκαν. Συμφωνούμε γενικά, αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Καταρχήν με τον Review Advisor. Η όλαφη Κομισιόν είναι υπέρ της δημιουργίας αυτής της θέσης που να επιβλέπει κατά πόσον υπάρχει νομιμότητα της κάθε έρευνας της Όλαφ. Είναι τόσο πολύ υπέρ μάλιστα, ώστε ήδη στην ουσία υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία. Ήδη δηλαδή βρίσκεται αυτή η πρόταση στην τροποποίηση της Κομισιόν του άρθρου 7β, όπου η εγγύηση της ανεξαρτησίας του Review Advisor αναφέρεται ρητά. Άρα συμφωνούμε όλοι επ' αυτού. Η μόνη διαφορά, η λεπτομέρεια όπου υπάρχει κάποια διαφορά κατανοητή είναι στο πρακτικό οργανωτικό θέμα. Δηλαδή αν το πρόσωπο αυτό πρέπει να διοριστεί μιας διαπαντός να έχει ένα γραφείο με έναν βοηθό και μια γραμματέα και να κάνει μόνο αυτό ή εάν οριστεί ή ορίζεται όποτε χρειάζεται. Αυτό εσείς θα το αποφασίσετε. Είναι οργανωτικό θέμα. Αλλά να σας δώσω δύο πληροφορίες. Πρώτον, τα τελευταία χρόνια το πολύ πέντε περιπτώσεις υπήρξαν όπου μπορεί να χρειαζόταν review advisor. Πέντε περιπτώσεις το χρόνο και κανονικά λιγότερο. Άρα μια μόνιμη τέτοια θέση θα σημαίνει ότι τον περισσότερο χρόνο δεν θα κάνουν τίποτα όσοι έχουν αυτή τη μόνιμη θέση. Αυτό δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή γιατί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά πρέπει να περικόψουν και τους ανθρώπινους και τους χρηματικούς τους πόρους. Αν τώρα μου λέτε ότι χρειάζονται περισσότερες, γρηγορότερες, καλύτερες έρευνες αλλά με περιορισμό των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων δεν μπορώ ταυτόχρονα μερικούς να τους βάλω να κάνουν μόνο τη δουλειά του Review Advisor Δεν γίνονται αυτά και τα δύο. Ή θα μου δώσετε περισσότερους πόρους ή δεν θα είναι μόνιμη αυτή η θέση. Τέλος πάντων αυτό είναι οργανωτική λεπτομέρεια. Γιατί όλοι μας θέλουν να υπάρχει review advisor ανεξάρτητος. Είναι λοιπόν θέμα οργάνωσης. Τουλάχιστον συμφωνούμε επί της ουσίας. Για την Επιτροπή Επιτήρησης, η κυρία Γιάλα μου Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Διότι πιστεύω και εγώ ότι μια τέτοια, αυτή η Επιτροπή θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα όπως ακριβώς είπατε να είναι πιο ορατή κλπ. Εσείς όμως πρέπει να επιλέξετε εκεί τους καταλληλότερους. Εγώ δεν έχω κανένα ρόλο να παίξω σε αυτό. Το Κοινοβούλιο όμως θα, και η Κομισιόν με το Συμβούλιο θα τα αποφασίσουν. Εγώ απλώς θα ήθελα όντως να υπάρχουν γνωστοί και πεπειραμένοι άνθρωποι σε αυτή την Επιτροπή. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Και ελπίζω να μπορέσετε να επιλέξετε τέτοιους κατάλληλους ανθρώπους. Αλλά Επιτρέψτε μου να μιλήσω και για το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Επιτήρησης, όπως είπατε όλοι και συμφωνώ και εγώ, εγγυάται την ανεξαρτησία της Όλαφ και του Γενικού της Διευθυντή. Επομένως, οι γνωμοδοτήσεις της δεν δίνονται μόνο στην ίδια την Όλαφ, αλλά και στα άλλα θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή Επιτήρησης πρόσφατα γνωμοδότησε για την υπόθεση Όλαφ Κοινοβούλιο και είπε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτά που είχε κάνει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Επιτήρησης αυτό το δήλωσε ακριβώς για να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της υπηρεσίας. Η ανεξαρτησία της Όλαφ λοιπόν δεν σημαίνει μόνο να ελέγχουμε τι κάνει η Όλαφ αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα. Ο καθένας πρέπει τουλάχιστον να ακούσει αυτές τις συστάσεις της Επιτροπής Επιτήρησης των Κατογνωμοδοτήσεών της. Τώρα ο αναπληρωματικός, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής. Εδώ ίσως υπάρξει μια παρεξήγηση. Κανείς δεν είπε να οριστεί αναπληρωτής γενικός διευθυντής. Και συμφωνώ με τον κύριο Γκάγερ, αν τον κατάλαβα καλά, ότι δεν χρειάζεται να οριστεί ένας αναπληρωτής γενικός διευθυντής. Και για τους λόγους που είπα πριν, την έλλειψη πόρων. Αλλά όχι μόνο. Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για το 12α λέει να υπάρξουν ορισμένοι κανόνες για την αναπλήρωση του Γενικού Διευθυντή, όχι για μόνιμη θέση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Για την περίπτωση που χρειάζεται να λείψει ο Γενικός Διευθυντής ή είναι σε άδεια ή έχει αρρωστήσει κλπ. Και λέει ότι γενικά στην Επιτροπή, στην Κομισιόν, ο κανόνας που ισχύει είναι όποιος έχει περισσότερη αρχαιότητα να παίζει αυτόν τον ρόλο όποτε χρειαστεί. Και αν ο Γενικός Διευθυντής θέλει να αλλάξει ο κανόνας αυτός, τότε να πρέπει να, να διαβουλευθεί με την Επιτροπή Επιτήρησης. Αν τώρα εσείς νομίζετε ότι στην περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής φύγει διακοπές και θέλει να παρακάμψει το γενικό κανόνα της αρχαιότητος που ισχύει στην Κομισιόν και για να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων διευθυντών που να μην είναι το αρχαιότερο μέλος δηλαδή, πρέπει να ρωτήσει την Επιτροπή Επιτήρησης και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, γιατί «Ε, πράγματα είναι αυτά. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύει πάντοτε ο απλούστερος κανόνας, δηλαδή του αρχαιότερου. Δεν μπορεί να διαβουλεύεται κανείς με τέσσερα όργανα για να πάει ο Γενικός Διευθυντής δύο εβδομάδες διακοπές ή για να αρρωστήσει για μερικές εβδομάδες προσωρινά για να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων ποιος θα με αναπληρώσει ας πούμε δεν, πρέπει, δεν είναι δυνατόν να πρέπει να ζητώ την άποψη τεσσάρων θεσμικών οργάνων είναι και αναξιοπρεπές αλλά τέλος πάντων αν μου το ζητήσετε δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα και αυτά λεπτομέρειες είναι γιατί επί της ουσίας πάλι συμφωνούμε. Και τελευταίο θέμα, για να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο τα κράτη-μέλη. Και από αυτού συμφωνούμε. Η δική μου στρατηγική είναι, αντί να παίζουν κάποιο ρόλο στο τέλος της έρευνας, να συμμετέχουν από την αρχή, κατά τη διάρκεια της έρευνας, για να μην χάνεται χρόνος όπως παρατηρείται πολλές φορές με τις διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Έτσι θα είναι και συντομότερες οι έρευνες. Αλλά πάλι αν μου το ζητήσετε, αν κάθε φορά πρέπει μια εθνική αρχή να περνάει από την Επιτροπή Επιτήρησης μία φορά το μήνα, δεν είναι λογικό κάτι τέτοιο. Αν πρέπει να απλοποιήσω και να επιταχύνω τις διαδικασίες και να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη από την αρχή, τότε αυτή η άδεια από την Επιτροπή Επιτήρησης είναι παρεμπόδιση, δεν είναι διευκόλυνση. Προς το παρόν αυτά είναι τα σχόλιά μου, αλλά είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Κύριε Γενική Διευθύντα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήρθε ο Ανατός Δικαστικός, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και ήδη ο συνεργάτης σας έκανε μια πρώτη εισήγηση άριστη για την εργασία σας. Μήπως θα επιθυμούσατε το λόγο για να συμπληρώσετε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα. Αυτό οφείλεται σε πρόβλημα κυκλοφοριακό. Νομίζω ότι η παρουσίαση του κ. Μπετραγκούκ που έγινε εκ μέρους ε, της Επιτροπής. Αυτήν την ε, εισήγηση στηρίζουμε και εμείς και σε αυτή τη φάση δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε. Θα ενημερωθώ για τη συζήτηση από τους συναντέλφους μου, ε, για αυτά που δεν άκουσα. Τώρα είμαι και εγώ εδώ και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο αυτού, αυτής της νομοθετικής πρότασης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Γκαλιά. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι θέλει να προσθέσει. Ακούσαμε τις διάφορες εισηγήσεις σχετικά με την πρόταση. Όχι, κανείς. Κανείς ο εισηγητή για να ολοκληρώσουμε. Η εισηγήτρια, συγγνώμη. Μήπω α, όχι, Μήπως το Συμβούλιο, ναι, αλλά δεν συνηθίζεται, δίστασα, ναι, μήπω ε, το Συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει την απόψή του. Καλό θα ήταν να μας λέει περισσότερα πράγματα το Συμβούλιο εδώ στην κοινοβουλευτική μας αυτή η Επιτροπή. Όχι, δεν επιθυμεί. Ε, επιφυλάσσεται ε, θέλει να εκφραστεί κατά τη διάρκεια των, διαπραγματεύσεων ασφαλώς. Λοιπόν, ο εισηγητής η εισηγήτρια μας να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση, ε, η ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους και να πω ότι αυτά τα οποία ελέγχθησαν ε, σήμερα το πρωί αφορούν την πεμπτουσία εκείνων ε, που θα συζητήσουμε κατά τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να προτείνω στους αδέλφους μία διαδικαστική πρόταση. Ε, δηλαδή έχουν οριστεί οι ε, σκιώδεις ηγητές και πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις των μόντων δυνατών. Βεβαίως πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιες λεπτομέρειες, ε, για κάποιες χρειαζόμαστε χρόνο, για άλλες λιγότερο. Ίσως αν περιμένουμε όλους το να βρούμε μια ημερομηνία με ταιριά σε όλους θα περάσει πολύ καιρό. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να δεχτείτε ότι ορισμένα πράγματα θα γίνονται από όλους μας αλλά υπάρχουν και κάποιες τεχνικές ημερομηνίες, τεχνικά ραντεβού για να ξεκαθαρίζουμε καταστάσεις και όσοι θέλουν μπορούν να έρχονται. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναλάβω εγώ να ε, ρυθμίσω αυτά τα τεχνικά ραντεβού ακόμα και αν δεν έρθουν όλοι γιατί αν πρέπει να περιμένουν να έρθουν όλοι, δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα, ε, προτείνω κάποιες ε, ημερομηνίες ε, καντιάκες της Προεδρίας και παρακαλώ να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις λεπτομέρειες, γιατί τα προβλήματα είναι οι λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όσο δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Έχω λοιπόν διατυπώσει 14 ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και με αυτέ θέλω να ξεκινήσω. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό το Συμβούλιο το οποίο στην πρότασή, της έχει, πρότασή του έχει παραμείνει πολύ κοντά σε αυτή την πρόταση Κομισιόν. Το Συμβούλιο λοιπόν ε, πρέπει να ενημερωθεί για το πού πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Αυτή είναι η δική μου πρόταση και ελπίζω να συμφωνούν και οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω μήπως ε, κάποια άλλη παρουσίαση. Όχι, τότε αυτή η πρόταση να συζητηθεί, αυτή η άριστη πρόταση να συζητηθεί ε, με τους συντονιστέ. Πάνω σε αυτό κάτι θέλετε να πείτε. Ναι, πρόεδρε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη διάθεση που δείχνει. Γνωρίζουμε τη δυνατότητά της εργασίας και θα ήθελα όμως να ζητήσω, να ζητήσω κάτι στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεών μας και σχετικά με τον κανονισμό κλπ. Να έχουμε συναντήσεις που να είναι αποτελεσματικές και όσο αφορά εναλλακτικά θέματα Εντάξει, το λέω έτσι με καλή διάθεση να πάρουμε θέσεις από πολιτικής πλευράς το θέμα αυτό της Όλαφ. Όλοι και οι συντονιστές έχετε αυτή τη ε, δυνατότητα να το θέσετε και να δούμε ακριβώς ε, ποια μπορούν να είναι τα σημεία κλειδιά τα οποία να απασχολούν τις συναντήσεις μας και όχι να το συζητάμε όπως το συζητάμε κανονικά σε μια επιτροπή αλλά να δούμε ακριβώς ε, θέματα και αποφάσεις σε σημαντικά πράγματα. Διαφορετικά έτσι συνεχείς επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις ε, και να βλέπουμε για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι συναντήσεις ε, τι γίνεται στο τέλος, ότι είναι αντιπαραγωγικό αυτό, δεν συναντή με τα υπόλοιπα, με το συμφέρον μας κλπ. και με όλα αυτά που θέτει και η συγκήτρια. Γι' αυτό σας παρακαλώ λοιπόν να το προετοιμάσουμε ώστε κάθε συνάντηση να μας ε, ωφελεί για να λύνουμε και όχι για να θέτουμε θέματα καινούρια. Ευχαριστώ την κυρία Γιάλα. Η πρόταση λοιπόν αυτή είναι να το συζητήσουμε αμέσως, για το, μάλλον να συζητήσουμε στις, με τους συντονιστές τι θα δοθεί σαν συνέχεια σε λίγο μετά από την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έτσι κλείνει εδώ το θέμα αυτό και να σας προτείνω το σημείο 6 Κανταράς, εκεί συνάντηση 16-18 Μαΐου, ο Μπαρθτάς πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, ε, ε, πρέπει να είναι αλλού και πριν να το συζητήσουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πώς έχουν γι' αυτό να το αναβάλουμε. Σήμερα το απόγευμα ανταλλαγή απόψεων σημοντακότατη για τα διάφορα πειθαρχικά θέματα και θα έχουμε και το διαμεσολαβητή, τον, κύριο Διαμαντούρο και τον Ζαν που είναι με ειδικέ γνώσεις ε, δικηγόρος για τα πειθαρχικά θέματα εδώ σε αυτή την αίθουσα λοιπόν την 2Q2 στις 3 η ώρα το απόγευμα θα συναντηθούμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε παρόντες γιατί είναι πολύ σημαντική σαν ακρόαση για το θεσμικό μας όργανο. Έτσι. Λοιπόν, ε, πέρα συνεδρίασης. 2Q2 σήμερα το απόγευμα. Τώρα παρακαλώ τους συντονιστές ε, μήπως θα μπορούσαμε να τα δούμε